Ε, μια αστική υπόθεση υπέρ του κυρίου Βίκτορ Μποστινόριου, η διαδικασία τη άρση ασυλία ολοκληρώθηκε. Τώρα, μετά από τι αποφάσει τη Επιτροπή ΕΚΟΝ να ξεκινήσει οι διαπραγματεύσει βάσει του άρθρου 69D, ε, δεν έλαβα κανένα ε, αίτημα και επομένω θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει μετά από την προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 69.4 παράγραφος 2 αποφασίστηκε να ξεκινήσουν διοργανικές διαπραγματεύσεις βάσει το, του άρθρου 69C παράγραφος 1 του κανονισμού. Οι νέες ε, σχέσεις οι οποίες καθορίζονται βρίσκονται στην ιστοσελίδα ε, της Ολομέλειας και οι τίτλοι θα δημοσιευθούν στα πρακτικά της Ολομέλειας. Βάσει του άρθρου 69C παράγραφος 2, ένας αριθμός ευρωβουλευτών ή μία περισσότερες πολιτικές ομάδες, οι οποίες θα πρέπει τουλάχιστον να βρίσκονται στο μέσο όρο, μπορούν να ζητήσουν γραπτός μέχρι τα μεσάνυχτα αύριο, 3η 29 Μαΐου, να ψηφιστεί η απόφαση για την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Εάν δεν υπάρχει σχετικό αίτημα, για ψηφοφορία στην Ολομέλεια για την απόφαση έναρξη διαπραγματεύσεων εντό αυτή τη προθεσμία, οι επιτροπή μπορεί να ξεκινήσουν τι διαπραγματεύσει. Η Επιτροπή Τραν διαβίωσε.